Er- Άρχεται η συνεδρίαση που διακόπη στις 24 Απριλίου Παρασκευή, περίοδο Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνεχίζεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από λίγες ημέρες είχαμε την επέτειο της πέμπτης